Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη καταρχά για αυτή την καθυστέρηση. Καθυστέρηση που οφειλόταν στην προετοιμασία του τριλόγου που θα έχουμε σήμερα το απόγευμα στις 4. Λοιπόν, έγκριση του σχεδίου ημερησίας διάταξης και Έχουμε τώρα το σημείο 7 που πρέπει να ψηφίσουμε, συνάδελφοι. Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό Έτο 2014, όλα τα τμήματα. Μετά την ε, ψηφοφορία για τις τροπολογίες θα πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεσή μας που συνοδεύει τις τροπολογίες. Η Ντάντσιλα θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την υποστήριξη και όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τις τροπολογίες στην έκθεση. Ευχαριστώ την κυρία Ντάντσιλα. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Α, η Μπρίτα ζητάει το λόγο. Με συγχωρείτε, δεν λειτουργεί η κάρτα ψηφοφοριών. Δεν λειτουργεί με κανένα τρόπο. Ας ψηφίσουμε με ανάταση χειρός. Ωραία. Ξεκινάμε με την παράγραφο 1. Υπέρ, παρακαλώ. Σηκώστε το χέρι σας. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Εγώ θα έλεγα ότι απορρίπτεται. Παράγραφος 3. Υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, θα εγκρίνεται, εγκρίνεται. 6. Λάιον. Υπέρ. κατά θα έλεγα ότι απορρίπτεται. Okay. Uh, Προφορική τροπολογία Ολενίτσακ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Τροπολογία 7. Στο Ιανόφ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 10. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 του Ελενίτσακ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 Γκάμπριελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα, πιστεύω. Τελική ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στην κυρία Ντάντσιλα. Πριν ασχοληθούμε με το επόμενο σημείο. Α, ο αντιπρόεδρος κύριος Μποβέ ζήτησε το λόγο. Ζωζέ. Συγγνώμη που ταράζω την μισή διάταξη, αλλά η πρόταση πρέπει να γίνει πρόταση και για την επόμενη άνοιξη, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν το 14 έτος οικογενειακής γεωργίας. Πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω να συμμετάσχει και αυτό στους εορτασμούς αυτούς και να οργανώσει μια εκδήλωση από την Επιτροπή Γεωργίας. Δεν υπάρχουν αγγλικά. Τώρα υπάρχουν. Ξαναρχίζω από την αρχή. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν το έτος 14 ως έτος της οικογενειακής γεωργίας. Θα οργανωθούν πολλές εκδηλώσεις παγκοσμίως για την οικογενειακή γεωργία και προτείνω η Επιτροπή Γεωργίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή, να αναλάβει μια πρωτοβουλία για την υπεράσπιση και προώθηση της οικογενειακής γεωργίας. Καλό θα ήταν νομίζω η Επιτροπή Γεωργίας να οργανώσει την εκδήλωση αυτή την Άνοιξη. Πριν όμως τον Απρίλιο, γιατί μετά θα είναι οι εκλογές, το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο δηλαδή να οργανώσουμε μια τέτοια εκδήλωση όπου να καλέσουμε προσώπους οργανώσεων διαφόρων τύπων γεωργίας και να στείλουμε επιστολή στη Γραμματεία στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου για να συμμετάσχουν όσοι θέλουν από το Κοινοβούλιο, όσοι συνάδελφοι θέλουν, γιατί νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό και ο Επίτροπος σε όλους να συμμετάσχει, ώστε να δείξει και η Ευρώπη ότι υποστηρίζει την οικογενειακή γεωργία. Σας κάνω την πρόταση προφορικά πριν στείλω μήνυμα και επιστολή, για να μπορέσουν και οι συντονιστές να το συζητήσουν. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο. Σημειώσαμε αυτά που μας είπε και τώρα θα έλεγα να ασχοληθούμε πρώτα με το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Είναι σημαντικό το σημείο αυτό γιατί θα πρέπει να ψηφίσουμε ούτως ή άλλως. Και θα ήθελα να παραμείνουν όλοι οι συνάδελφοι στην αίθουσα. Θα θυμόσαστε αγαπητοί συνάδελφοι, εκτός από τα μεταβατικά μέτρα για το 2014 που ο Άλμπερτ Έσσι είναι ο εισηγητής, η Επιτροπή τον Ιούλιο υπέβαλε μία πρόταση νομοθετικού προϊριοχωμένου για μεταβατικά μέτρα τα οποία ασχολούνται, έχουν να κάνουν με, με τον κανονισμό 1698 του 2005 για την ανάπτυξη της ε, υπαίθρου. Η μόνη διάταξη σε αυτή την πρόταση είναι μια παράταση της ισχύουσας παρέκκλησης για την χρήση ε, συγχρηματοδότησης ε, από τα κράτη-μέλη. Μετά από μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τους συντονιστές αυτό το θέμα, θεωρώ ότι το θέμα αυτό δεν, είναι, δεν δημιουργεί προβλήματα. Όμως η όλη διαδικασία είναι λίγο ε, περίπλοκη και θα πρέπει να υπάρξει μία διαδικασία συναπόφασης και αυτό μέσα από μία απλουστευμένη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 46. Παράλληλα όμως, όπως συμφωνήσαμε και με τους συντονιστές, ο κύριος Σέσε υπέβαλε και μία αντίστοιχη τροπολογία στην έκθεσή του που προτείνει αυτή η παράταση να συμπεριληφθεί στην πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Τέσσερις τροπολογίες, αν γίνουν δεκτές από το Συμβούλιο και υιοθετηθούν και στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απόσυρση για την πρόταση της ε, Κομισιόν. Επομένως, συνάδελφοι, προτείνω να υιοθετήσουμε αυτή την πρόταση με την απλουστευμένη διαδικασία χωρίς τροπολογίες, εφόσον το περιεχόμενο δεν ε, έχει καμία αρνητική συνέπεια. Βλέπω ότι ο κύριος Ντές ε, γνέφει καταφατικά, άρα εφόσον δεν υπάρχουν ε, ε, συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο, θα ήθελα να σας ζητήσω να ψηφίσουμε την πρότασή μου. Ποιος είναι υπέρ αυτή τη εφαρμογή απλοποιημένη διαδικασία, υπέρ, κατά Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ντέσε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Πάρα πολύ ωραία. Εάν ε, συμφωνείτε κι εσείς, μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, ε, που είναι η παρουσίαση του, από πλευράς του Μαωρίτσιο Μαρτίνα, που είναι υφυπουργό Γεωργικής Βιομηχανίας Τροφίμων και Δασικών Πολιτικών της Ιταλίας, σχετικά με την παγκόσμια έκθεση του 2015. Τροφή για τον πλανήτη ενέργεια πηγή ζωής. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους, όλους όσους είναι παρόντες ε, σε αυτή την ε, πρώτη παρουσίαση για την Διεθνή Έκθεση του 2015. Όπως ξέρετε θα έχει σαν ε, στόχο, αν θέλετε, σαν κύριο θέμα την τροφή. Βέβαια όλα αυτά έχουν αποκτήσει και άλλες διαστάσεις και θίγουν πολλές ευαισθησίες. Το θέμα της διατροφής είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον πλανήτη και εδώ συνδέονται και θέματα βιωσιμότητας του πλανήτη. Έχουν γίνει διάφορες αναλύσεις ε, μετά την άνοδο των τιμών το 2006 έδειξαν ε, ποια είναι τα προβλήματα, τα παγκόσμια προβλήματα για την διατροφική ε, ασφάλεια, για, για τον επισητισμό. Είναι περίπλοκα όλα τα στοιχεία τα οποία εμφανίζονται είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο, συνάδελφοι. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές ε, στην Επιτροπή μας και πάρα πολύ συχνά έχουμε υπογραμμίσει την σημασία που έχει να λάβουμε υπόψη μας αυτή την παγκόσμια πρόκληση που αποτελεί την επιστηστική ασφάλεια. Και όλο αυτό μέσα στα πλαίσια και του μεγάλου διαλόγου που είχαμε για την μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής σήμερα που μπορώ να ε, υποδεχτώ τον ε, Υφυπουργό, τον κύριο Μαρτίνα, που θα μας παρουσιάσει με κάποιες διαφάνειες ποιος, ε, είναι ο στόχος αυτής της διεθνούς έκθεσης που μας αφορά όλους, όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά όλη την, ε, όχι μόνο την Ιταλία αλλά όλη την Ευρώπη και νομίζω ότι ε, είναι και ένα φόρουμ μέσα από το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις. Ευχαριστώ ε, όλους, ε, όλη την αντιπροσωπεία της Ιταλίας που έχει έρθει εδώ και θα δώσω τον λόγο αμέσως στον Υπουργό, τον κύριο Μαρτίνα, μετά ξέρω ότι θα είναι και παρόντες ε, και συνάδελφοι από άλλες επιτροπές, θα τους δώσω το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο και στους συναδέλφους από την Επιτροπή Γεωργίας ε, και από τους συντονιστέ των πολιτικών ομάδων σε όσους ζητήσουν το λόγο βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο τον έχει ο Μαουρίτσιο Μαρτίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο, ευχαριστώ όλους σας την Επιτροπή για μας είναι μια μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση που είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε το έργο το οποίο έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα για, να, για αυτή την ε, διεθνή έκθεση του Μιλάνου του 2015. Θα ήθελα μέσα σε λίγα λεπτά να τονίσω την σημασία που έχει η απόφαση για να, να γίνει η έκθεση στο Μιλάνο, ε, ποια είναι τα αριθμητικά στοιχεία και μετά θα ασχοληθώ με κάποια σημαντικά στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα ε, της έκθεσης ε, για το 2015. Κυρίως και σε σχέση με αυτά που είπε και ο πρόεδρος Δεκάστρο. Μία πρώτη φωτογραφία να δείτε, ε, μία πρώτη παρουσίαση αν θέλετε, των αριθμητικών στοιχείων για την ε, ε, έκθεση του 2015 που θα λάβει χώρα στο Μιλάνο από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2015. Μέχρι στιγμής έχουμε εξασφαλίσει την συμμετοχή 132 χωρών ε, να λάβετε υπόψη σας ότι ο στόχος μας ήταν 130, τον ξεπεράσαμε το στόχο μας ε, δηλαδή και προβλέπουμε ότι θα, τις επόμενες εβδομάδες ε, θα εξασφαλίσουμε και άλλες συμμετοχές για, αυτή, αυτό το μεγάλο ραντεβού. 60 χώρες εκ των οποίων των οποίων θα έχουν 132 χώρες τα δικά τους ε, περίπτερα. Ε, στην Σανγκάη βέβαια από αυτές τις 132 χώρες οι 60 θα έχουν τα δικά τους ε, περίπτερα. Στη Σανγκάη για για να καταλάβετε την Πώ ε, γίνονται τα πράγματα. Έχετε ένα μέτρο σύγκριση. Στη Σανγκάη είχαμε 40 περίπτωρα. Και ε, ελπίζουμε ότι θα μας επισκεφθούν 20 εκατομμύρια ε, επισκέπτες. Ο χώρος της έκθεσης είναι ένα εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Η επένδυση από πλευράς της Ιταλίας είναι 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, υπάρχει και επένδυση ε, από τις συμμετέχουσες χώρες βέβαια που ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο περίπου και αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ που η οργάνωση έχει εξασφαλίσει από ιδιώτες επενδυτές. Βλέπετε εδώ ε, στην διαφάνεια αυτή τις διάφορε διάφορες ε, ε, σημαίες των ε, συμμετεχουσών χωρών. 132 χώρες όπως είπαμε συμμετέχουν και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι ήδη έχουμε εξασφαλίσει μια μεγάλη συμμετοχή χωρών από την Ασία, από την Αφρική και σε αυτό το πλαίσιο πάντα λέμε ότι το 97% της, του πληθυσμού ε, της Ασίας θα εκπροσωπείται μέσω των κρατών του στην ε, έκθεσή μας. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό γεγονός ε, και είναι και στρατηγική σημασία, θα έλεγα, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροφή για τον πλανήτη, η ενέργεια πηγή ζωή, όπως είπε και ο πρόεδρος Ντεκάστρο, αποτελεί την βασική μας πρόταση, τον πυρήνα της πρότασής μας. Όπως ξέρετε, καλή, καλύτερα από μένα κιόλα, θα πρέπει να συζητήσουμε με όλο τον πλανήτη τα νέα σύνορα ε, για την διατροφή, τις ε, νέες πολιτικές ε, για την βιωσιμότητα. Θα πρέπει να δούμε κιόλας εδώ κάποια εντυπωσιακά αριθμητικά στοιχεία, τα οποία τα γνωρίζουμε, αλλά θα πρέπει να τα προβάλλουμε και στην ευρωπαϊκή και διεθνή κοινή γνώμη να υπενθυμίσουμε απλώς και μόνο και να σκεφτούμε κάποια εντυπωσιακά στοιχεία. 800 εκατομμύρια ε, άτομα υποσυτίζονται, 1,5 δισεκατομμύρια είναι παχύσαρκοι, ένα στα τρία άτομα έχουν προβλήματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα διατροφής και σε κάθε υποσυτισμένο άτομο έχουν, ε, αντιστοιχούν δύο υπέρβαροι, δύο παχύσαρκοι μάλλον και ο βασικός στόχος είναι να ψάξουμε να βρούμε στο Μιλάνο μια νέα ισορροπία ε, ανάμεσα στην παραγωγή και στην ε, κατανάλωση των τροφών μέσα στα πλαίσια μιας ανανεωμένης σχέσης με το περιβάλλον. Στοιχεία που γνωρίζετε βέβαια και τα, τα συζητάει η Επιτροπή σε όλα αυτά τα θέματα και τα θέματα προσφοράς, ζήτησης, ε, την ανισορροπία που υπάρχει ανάμεσα στην ε, προσφορά και στην ζήτηση και ακριβώς όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν το εύρος και το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε. Επομένως, η, η διατροφή, ο επισητισμός αν θέλετε, είναι το μεγάλο θέμα, η μεγάλη πρόκληση που θα αντιμετωπίζουμε και τώρα και στο μέλλον. Στο 2015 θέλουμε να συζητήσουμε κάποια βασικά θέματα που μας αφορούν και όλους και που συζητούνται και σε κάποια θεσμικά όργανα. Το ένα είναι αυτή η κούρσα για να εξασφαλίσουμε ε, την, την γη, ε, κράτη, ε, οικονομικοί οργανισμοί προσπαθούν να εξασφαλίσουν γεωργικούς πόρους. Η η διακύμανση που, που παρουσιάζει η αγορά όσον αφορά τις τιμές και που πλήττει ε, τους πληθυσμούς, ε, τους πιο φτωχούς πληθυσμούς, ε, οι κανόνες στην διεθνή αγορά έχουμε μπει σε αυτή την εποχή του ανάποδου προστατευτισμού όπου εξάγουμε τροφή μεν και εξάγουμε ταυτόχρονα και πληθωρισμό. Επομένως, ε, πρέπει να υπάρχει, ε, ε, θεωρούμε ότι η έκθεση ε, θα αποτελέσει ένα φόρουμ έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε το μείζον θέμα της σχέσης γεωργίας και περιβάλλοντος, τα θέματα βιωσιμότητας και ανταγωνισμού, μια νέα σχέση ανάμεσα στην γεωργία, την τροφή και την ευημερία, διότι η διατροφή προσφέρει στην ευημερία προφανώς των πληθυσμών. Ένα άλλο θέμα είναι η διατροφή και οι καινοτομίες, έρευνα γνώσης, μεταφορά ε, γνώσεων ε, με βάση την ε, επιστημιστική ασφάλεια και την ασφάλεια των τροφίμων και μετά έναν βασικό στόχο, έναν μείζωνα στόχο που είναι ε, το θέμα της διατροφής να αποτελέσει ένα κομμάτι των μεγάλων, των, μεγάλων πολιτικών, των πολιτικών μάλλον που συζητούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, δηλαδή να συζητείτε το θέμα ε, σε φόρα όπως το G8 ή το G20 εκεί να συζητώνται πώς δημιουργούνται νέες πολιτικές το βασικό επιχείρημα που επέτρεψε στο Μιλάνο να κερδίσει την έκθεση ε, περιλαμβάνει τέσσερα βασικά θέματα. Επιστηστική ασφάλεια, ασφάλεια τροφίμων, η, η βιωσιμότητα και ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης πιο ισορροπημένο και μετά σχέση ανάμεσα στην τροφή, την ειρήνη και τη γνώση. Αυτό το στρατηγικό έγγραφο που μας επέτρεψε να εξασφαλίσουμε την ε, ε, την ε, έκθεση μας επιτρέπει να ε, διαβουλευόμεθα και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2015 και πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συντάξουμε έναν ηθικό κώδικα εναντίον όλων των όλης να έχουμε μια μοιρασμένη ε, δέσμευση για να περιορίσουμε όλες τις ε, πολιτικές ε, τις κερδοσκοπικές και ε, επίσης θα πρέπει να υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διατροφής και υπάρχει και το πρόγραμμα του ΟΗΕ ταυτόχρονα ε, παράλληλα, το οποίο ολοκληρώνει το 2015. Επομένως θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τα αντιμετωπίσουμε σφαιρικά, έτσι ώστε να προωθήσουμε κάποια θέματα τα οποία δεν τα είχαμε ε, συζητήσει επαρκώς μέχρι τώρα. Βλέπετε εδώ ποια είναι η περιοχή όπου θα λάβει χώρα η έκθεση. Είναι μεγάλη περιοχή προφανώς ε, και είναι και δύσκολο να ε, εξασφαλίσουμε την υποδοχή που θα θέλαμε για όλους τους επισκέπτες μας και θα ήθελα να αναφερθώ πριν κλείσω στην καινοτομία ε, που θέλουμε να εξασφαλίσουμε σε αυτή την έκθεση του 2015, γιατί ε, εδώ παρουσιάζουμε μια νέα μορφή στις ε, διεθνείς εκθέσεις. Έχουμε δημιουργήσει διάφορα clusters, δηλαδή δεν ε, έχουμε μόνο αυτόνομη παρουσία κρατών με τα δικά τους περίπτερα, αλλά έχουμε υποβάλει μια πρόταση όπου θα, έχουμε, θα υπάρχουν εννέα, νέα θεματικά κλάστερ για κάθε συγκεκριμένα θέματα για κάθε ε, διατροφική αλυσίδα κτλ. Ε, θέλουμε να υπάρχουν θα υπάρχει κάθε κράτος να παρουσιάζει την δική του ε, γεωργική παραγωγή τέλο πάντων. Δηλαδή μέσα από τον καφέ, το ρύζι, τα μπαχαρικά, τα δημητριακά, τα προκυπευτικά κτλ. Θα κάνουμε μια αντιπαράθεση σε επίπεδο project ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει δηλαδή τα κράτη-μέλη αυτόνομα να παρουσιάζουν την δική τους εικόνα, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούν ε, και με τα άλλα κράτη και να υπάρχει μια συνδυασμένη παρουσίαση με βάση κάποιες ε, αυτά τα, τα εννέα κλάστερς. Και ελπίζουμε ότι αυτό το παράδειγμά μας θα το ακολουθήσουν και μελλοντικέ ε, εκθέσεις. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω, να πω ποια είναι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. το 2013, τον Μάρτιο, έγινε μία ανακοίνωση της Κομισιόν που παρουσιάζει την ε, παρουσία της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής στην Παγκόσμια Έκθεση. Καταρχάς θα υπάρχει παρουσία και χωροταξικά κιόλα μπροστά από το Παλάτσο Ιτάλια, στην καρδιά δηλαδή τη Παγκόσμια Έκθεση, σε παρουσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή ρυθμίζονται τελευταίε λεπτομέρειε οργανωτικέ, αλλά είναι ένα γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ε, παρούσα και σε περίοπτη θέση, θα έλεγα, στην έκθεση του 2015. Επίση, ορίστηκε ένας επίτροπος ε, ο Δόκτωρ Ντέιβιτ Wilkinson, ο υπεύθυνο και ένας αντιπρόεδρος, ο Τζαν Κάρλο Καράτη, με, τον, με τους οποίους συνεργαζόμαστε για να ε, επιλύσουμε κάποια λειτουργικά θέματα και ε, πιστεύω ότι η, έκθεση αυτή του 2015 πρέπει να γίνει μια ουσιαστική, μια βασική έκθεση που θα επηρεάσει και τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή σε όλα αυτά τα θέματα, σε παγκόσμια, παγκόσμια σκηνή. Και είναι απόλυτα διαθέσιμη και η Ιταλική κυβέρνηση αλλά και οι οργανωτές να συνεργαστούν μέχρι το 2015 έτσι ώστε να βελτιώσουμε ένα όλο πρόγραμμα συναντήσεων, ε, project, να γίνει μια προσέγγιση δηλαδή με, το, με την Expo 2015 έτσι ώστε η έκθεση αυτή να γίνει μια παγκόσμια ευρωπαϊκή έκθεση. Και θεωρούμε ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει να είναι μια πραγματική, η πρώτη πραγματική έκθεση με ευρωπαϊκό χαρακτήρα, διότι πιστεύω ότι θα έχει και βασικό θέμα, ε, θα έχει βασικό ε, συνδρομή, θα γίνει βασική συνδρομή και στις σχέσεις μας ε, σε διεθνές επίπεδο. Πιστεύω ότι όλοι είναι διαθέσιμοι να κάνουν αυτό το ποιοτικό άλμα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής ε, για αυτή την πρώτη συνάντηση, την οποία θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο βήμα και θα ακολουθήσουν και άλλα έτσι ώστε να μπούμε σε περισσότερες Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαρτίνα. Συνάδελφοι, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας στα πλαίσια της έκθεσης 2015 ε, στο Μιλάνο «Τροφή για τον πλανήτη ενέργεια πηγή ζωής» ε, να μην αποτελέσει απλώς ένα βήμα συζήτησης, αλλά να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης αυτής που θα έχει ένα παγκόσμιο χαρακτήρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ε, ε, παρέμβαση του Ιταλού Υπουργού. Θα ήθελα να ακούσω τώρα τις δικές σας ε, παρατηρήσεις, ξεκινώντας από τους συναδέλφους των άλλων επιτροπών. Ποιος, θα, ζητάει το λόγο? Η Πατρίτσια Τόλια, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας ενέργειας και έρευνας. έρευνας. Επιτροπή Ήτρε. Και μετά στους συναδέλφους που θα γνωστοποιήσουν στην γραμματεία την υποχρέωσή τους, την ε, θέλησή τους να μιλήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να, να καλωσορίσω και τον εκπρόσωπο της τελικής Κυβέρνησης, τον κύριο Μαουρίτσιο Μαρτίνα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ντεκάστρο, γιατί σαν ε, Επιτροπή Βιομηχανίας ε, συζητάμε τα θέματα αυτά και συνεργαζόμαστε και πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό να αντιμετωπίζουμε όλοι τα θέματα αυτά που μας απασχολούν τώρα σαν αντικείμενο συνεργασίες ανάμεσα σε όλες τις επιτροπές. Ε, πιστεύω ότι η εκδήλωση αυτή, η έκθεση δηλαδή, αυτή η συγκεκριμένη έκθεση που μας παρουσιάστηκε είναι μια εξωτερική, εξαιρετική συγγνώμη, εκδήλωση και ιδιαίτερα καινοτόμος, κυρίως όσον αφορά την ε, οργάνωση αλλά και αυτό το άνοιγμα στην Ευρώπη. Ε, οι διεθνείς ε, εκθέσεις στο παρελθόν Ε, ήταν μια παρουσίαση απλώς ε, των διαφόρων κρατών που συμμετείχαν. Εδώ, σε αυτή την έκθεση, πιστεύω ότι ε, η Ιταλία ζητάει από, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάσει την, μια καινούργια εικόνα. Και η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απλώς και μόνο το, η παρουσία ενός δικού της ε, περιπτέρου, αλλά ε, παρουσιάζονται, παρουσιάζεται οι, οι Ευρωπαίοι πολίτες και ε, μέσα από τους Ευρωπαίους πολίτες ε, θα υπάρξει και, αυτός, ε, και αυτή η συνεργασία και αυτή η συνδιαλλαγή και με τους πολίτες των άλλων χωρών που θα είναι παρόντες, παρούσες, συγγνώμη, παραδείγματος χάρη, χώρες και με τις οποίες έχουμε και πολλές επαφές. Επομένως θα είμαστε και εμείς πρωταγωνιστές σαν κοινοβούλιο. Ε, αυτό το θέμα της ε, διατροφής είναι ένα ουσιαστικό θέμα γιατί είναι παγκόσμια βιωσιμότητα παράλληλα με την ε, ενέργεια και άλλα θέματα γιατί η διατροφή τι σημαίνει γεωργία και νερό. Επίσης υπάρχουν και, είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα άλλα προγράμματα τα ερευνητικά. και εμάς μας, απασχολεί, μας απασχολούν επίσης και οι προκλήσεις της χιλιετίας, στις διάφορες προκλήσεις για το κλίμα, για την καινοτομία, για την ε, κοινωνική καινοτομία κτλ. Υπάρχει και η διατροφή. Επομένως υπάρχει μια ολόκληρη, ε, ένα ολόκληρο κεφάλαιο που ανοίγει τώρα για ε, δουλειά και, και εδώ μπαίνει και η έκθεση του 2015. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η τροφή είναι μια μεγάλη πρόκληση και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας θα συζητηθεί το θέμα της διατροφής με όλες ε, τις ε, συνιστώσεις, μεταφορές, ε, οργάνωση, οτιδήποτε αφορά την διατροφή και την βιομηχανία. Επομένως είναι δύο θέματα πάρα πολύ σημαντικά και η ΕΞΠΟ θα πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει καταλήτη. Μια τελευταία παρατήρηση και ολοκληρώνω mm. στην ε, πιστεύω ότι στην, στα, σε επίπεδο παγκόσμιας συνεργασίας ε, η έκθεση θα αποτελέσει ένα βήμα. Ξέρετε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά θέματα και για τα ε, καύσιμα αγροτικής προέλευσης ο κύριος Μαρτίνα αναφέρθηκε και στο θέμα της τροφής ειρήνης και της ειρήνης. Και εδώ θα έβαζα και εγώ Και ένα άλλο θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ στην Ευρώπη, σε όλες τις επιτροπές, ε, είναι κάτι το οποίο ε, απασχολεί όλες τις επιχειρήσεις, ε, τις ευρωπαϊκές, και αφορά το ότι προσπαθούν κράτη, οργανισμοί κτλ. να εξασφαλίσουν γη. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι από το Μιλάνο να υπάρξουν, να βγουν κάποιες, ε, ε, κάποιοι ελάχιστοι κανόνες όσον αφορά την μεταφορά κατοχής γεών. Γιατί υπάρχουν τεράστιες περιοχές τις οποίες τις έχουν ε, αρπάξει αν θέλετε διάφορες πολυεθνικές εταιρείες κτλ. Και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Δηλαδή πιστεύουμε ότι από το Μιλάνο μπορεί να βγει μια, ελάχιστη αν θέλετε νομοθεσία ή πρόταση για, νομοθετική ρύθμιση αυτών των ε, μεταφορών των γεών. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλες παρεμβάσεις ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Τόστμαν και μετά στον Άντριου. Ehm, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα θέματα αυτά της έκθεσης. Μία πάρα πολύ σύντομη ερώτηση. Είπατε ότι παράλληλα με την έκθεση, ας πούμε, με την παρουσίαση των διαφόρων θεμάτων, θα γίνουν και, και διαλέξεις και σεμινάρια ε, για θέματα που ε, συζητάει για αυτή τη στιγμή και η Επιτροπή μας και είπατε ότι θα υπάρξει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπετε και μία συνεργασία και με το Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή μας δηλαδή και θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι για κάποια θέματα τα οποία θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της Expo 2015 η δική μας επιτροπή θα μπορούσε να συμμετέχει. Ε, έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο, υπάρχει κάποια συνεργασία με τις ε, υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ρώμη, στο Μιλάνο για να προετοιμαστεί αυτή η παρουσία. Έρικ και μετά ο Μαγκίνες. <coughs> Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μαωρίτσιο Μαρτίνα για την ποιότητα της παρουσίασης και ε, για το πόσο σκόπιμο είναι το πρόγραμμα που μας προτείνεται. Όλα τα θέματα αυτά, όλα τα θέματα που μας απασχολούν αναφέρθηκαν. Φυσικά πρέπει ακόμη να γίνει δουλειά για να γίνει πιο κατανοητό το θέμα. Εμείς Οπωσδήποτε θα συμμετάσχουμε σε αυτή την προσπάθεια της παγκόσμιας έκθεσης. Το θέμα της ε, παραγωγής ε, μας απασχόλησε ε, και της αλλαγής του τρόπου παραγωγής μας απασχόλησε σε όλη την προσπάθεια μεταρρύθμισης της κοινή γεωρικής πολιτικής. Πώς θα παράγουμε, πώς θα καταναλώνουμε διαφορετικά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε στην τύχη όλα αυτά τα θέματα και πέρα από το θέμα του μάρκετινγκ της εμπορίας, γιατί τίθεται και αυτό το θέμα, είναι βασικό να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους εμπλεκομένους για θέματα επισητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι θεμελιώδες θέμα. Και είμαι πεπισμένος, Πρόεδρε, ότι πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία που μας παρουσιάστηκε. Κάθε τμήμα της προσπάθειας αυτής συνδέεται άρρηκτα με τα θέματα που μας απασχολούν. Είναι θέμα όχι μόνο του αμέσου μέλλοντος, αλλά και του μακροπροθέσμου. Και τα θέματα που τίθενται είναι ουσιώδη για την ε, συνολική προσπάθεια θεωρητικής αναζήτησης πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτά που είπε ο κύριος Μαρτίνα είναι πολύ σκόπιμα και εμείς ως Επιτροπή πρέπει τα θέματα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ, Έρικ. Μαγκίνες. Και μετά σε κυρίες και Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτήν την ε, θαυμάσια παρουσίαση. Θα καλύψετε τόσο πολλά θέματα. Άρα δεν μπορούμε να καταλήξουμε ήδη σε συμπεράσματα. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα, αλλά σας συγχαίρω για τη δομή των προτάσεών σας. Τώρα, για τη γεωργία. Ένα βασικό θέμα. Ε, αναφερθήκατε μάλιστα στο θέμα της ε, οικογενειακής Το θέμα είναι το εισόδημα της οικογενειακής γεωργίας. Και θα έπρεπε και εμείς να το τονίσουμε περισσότερο. Το αναφέραμε στο θέμα της, ε, των ιδιαίτερων διακυμάνσεων τιμών και για θέματα λοιπόν ε, ευστάθεια στην αγορά. Αλλά θα διαπιστώσουμε ότι παρά την συμβολή της κοινή γεωργικής πολιτικής το εισόδημα των γεωργών είναι χαμηλότερο από το μέσο εισόδημα των εργαζομένων στην Ένωση. Άρα πρέπει να το εξετάσουμε, να το συζητήσουμε περαιτέρω. Όχι μόνο ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι τιμές που λαμβάνουν για τα προϊόντα του είναι επαρκεί, αλλά να είναι λογικέ και οι τιμέ των εισρωών των γεωργών. Και αυτό είναι θεμελιώδες και έχει και περιβαλλοντική επίπτωση. Για την προσπάθεια αρπαγής γεών, land grabbing, το συζητήσαμε και σε άλλες επιτροπές. Κανείς δεν έχει προτείνει λύση. Γιατί ίσω δεν υπάρχει εύκολη λύση. Ακόμη και εντό τη Ευρώπη. πρέπει να μιλήσουμε για την χρήση των γεών. Αλλά σε χώρες όπως η Ιρλανδία, ξέρετε, το δικαίωμα ιδιοκτησίας ε, είναι θεμελιώδες, είναι στο Σύνταγμα. Είναι λοιπόν πολύ λεπτά τα θέματα αυτά. Και αυτό που οι αρμόδιοι για τη γεωργία θεωρούν καλό, πολλές φορές ε, απορρίπτεται από τους ε, περιβαλλοντολόγους. Το θέμα αυτό μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις, διενέξεις, αλλά και συμμαχίες. Τα απόβλητα. Φυσικά θέλουμε να τα αποφύγουμε. Αλλά αν μειώσουμε τα απόβλητα, δεν θα έχει επίπτωση αυτό στην τιμή των γεωργικών προϊόντων. Αρνητική επίπτωση. Βεβαίως για λόγους βιωσιμότητας ε, δεν βλέπουμε να πετάμε τρόφιμα. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ μείωσης ε, της σπατάλησης τροφίμων και άλλων πλευρών του προβλήματος. Θα προτιμούσα να τα έχουμε συνδέσει περισσότερο, να μπορούμε να τα συνδέσουμε, να βρούμε συνδυασμένη λύση. Πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο. Και από τις επισκέψεις μου σε χώρες που δεν έχουν ε, πολύ αναπτυγμένη γεωργία, θεωρώ ότι πρέπει να επιτρέψουμε στον αναπτυσσόμενο κόσμο να κάνει καλύτερη χρήση της γης, να αναπτύξει βιώσιμη γεωργία, ούτως ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξή τους. Και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε σε αυτήν την έκθεση και να δούμε και τον ρόλο των γυναικών σε αυτό. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, στι αναπτυσσόμενε χώρε, παίζουν ε, θεμελιώδη ρόλο στη γεωργία. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εντυπωσιακή προσπάθειά σα ε, Με δέος την ε, εξετάζω και ελπίζω να συμμετάσχουν και άλλε χώρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μάριοτ. Ο Αντιπρόεδρος Σεκερίεσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε και ο Υφυπουργό, θα τεθεί εδώ και στην έκθεση το θέμα του νερού των δάτων, αλλά θα ήθελα να το τονίσω κι εγώ. Γιατί στο άμεσο μέλλον το νερό θα αποτελέσει πολύ κρίσιμο πρόβλημα για την ανάπτυξη. Όσο συντομότερα λύσουμε το θέμα του νερού, μάλλον τα ενεργειακά προβλήματα είναι πιο εύκολο να λυθούν παρά το πρόβλημα του νερού. Επομένως δεν πρέπει να το αγνοήσουμε και στην έκθεση αυτή. Αν δεν θέλει κανείς άλλος να μιλήσει, να δώσω το λόγο στον Αντώνιο Παντζέρη που τον φιλοξενούμε σήμερα. Είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας μας για σχέσεις με τις χώρες Μαγκρέμ. Ευχαριστώ. Δύσκολο να, να καταλάβουμε τη σχέση έχει τώρα η εξωτερική πολιτική με το Μαγκρέμ ε, με τα θέματα αλλά για τις χώρες Μαγκρέμπ, με τις οποίες ασχολείται την προσωπία μου, είναι πολύ σχετική η Γεωργία και αυτή η έκθεση Μιλάνου 2015 γιατί έχει να κάνει με τον επιστημισμό, την ε, έρευνα, τις υποδομές. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Ε, είναι σημαντικά βέβαια και για την Ευρώπη στο σύνολό της το θέμα της επιστημιστικής ασφάλειας και ισορροπίας. Και αυτό το θέμα έχει μία επίπτωση. Και βεβαίως σχετίζεται και το θέμα της χρήσης υδάτων που έχει να κάνει φυσικά με την γεωργία. Και σημειώνω ότι στον πλανήτη μας υπάρχουν πολλές περιοχές όπου συνολικά η γεωστρατηγική ε, πολιτική και οι γεωστρατηγικές ε, απόψεις σχετίζονται πολύ με το θέμα των τροφίμων και των υδάτων και αυτά προκαλούν, όπως ξέρετε, και τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμών. Η μετανάστευση δεν οφείλεται μόνο σε πολέμους, εμφυλίους κτλ. Ο κύριος λόγος μετακίνησης πληθυσμών έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και τις δυνατότητες που έχουν να επιβιώσουν οι πληθυσμοί στις χώρες που βρίσκονται. Παίζουν ρόλο λοιπόν ε, και στα μεταναστευτικά κύματα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι παράλληλα με το θέμα της παραγωγής, της έρευνας και του μέλλοντος της αγροεπιστητικής, της γεωργικο-επιστητικής βιομηχανίας ή συνδέονται και τα θέματα, με παράλληλα με τα θέματα αυτά πρέπει να δούμε και τη σχέση με την εξωτερική πολιτική που έχει και θα ήταν σκόπιμο να το συζητήσουμε στην έκθεση αυτή του Μιλάνου του 2015. Να εξετάσουμε δηλαδή πώς θα συζητήσουμε το πρωτόκολλο του Κιώτο ή το κατά πόσο έχει εφαρμοστεί στο Μιλάνο ακριβώς το 2015. Ίσως ήταν μια καλή ευκαιρία να καθορίσουμε μια νέα προσέγγιση μέσω της συμβολής και των χωρών που θα συμμετέχουν ακριβώς στην έκθεση. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Βεβαίως τα θέματα αυτά δεν είναι απλά. Η γη μας αντιμετωπίζει τεράστιες δυσχέρειες και θα ήταν χρήσιμο να τη συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, η πρόκληση είναι μεγάλη και απαιτεί μια συνεργασία όλων μας και είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο από τη δική μας Επιτροπή, από, αλλά και από άλλο το Κοινοβούλιο, η συμμετοχή σε αυτή την, και η παρουσία σε αυτή την ε, μεγάλη πρόκληση είναι σίγουρη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Μαρτίνα για να ολοκληρώσει την παρουσίασή του και μετά θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο, όλους σας. Ε, πραγματικά θεωρώ πολύ θετικές ε, τις παρατηρήσεις ε, που κάνατε. Πραγματικά μας ενθαρρύνουν κυρίως όσον αφορά την, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων ε, που θα, που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκθεση αυτή και μέσα στα πλαίσια της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπα... η Επιτροπή σας μπορεί να παίξει ένα εξέχοντα ρόλο και θα πρέπει ε, ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανώσει την παρουσία της, αυτό το εξάμεινο της έκθεσης. Εμείς ε, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε και η Επιτροπή να είναι πρωταγωνίστρια ε, στις δραστηριότητες. Κάποια θέματα απλώς εγώ έθιξα στην παρουσία μου και ε, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικά, π.χ. το εισόδημα που, το θέμα του νερού. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού της έκθεσης να μπορέσουμε να οργανώσουμε κάποιες συναντήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν να συγκεκριμενοποιήσουν κάποιες λύσεις, κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και πιστεύω πραγματικά ότι θα πρέπει να εργαστούμε μέχρι την 1η Μαΐου του 2015 σε όλα τα φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε την το ρόλο της έκθεσης αυτής. Ε, πιστεύω ότι αυτή η έκθεση στην καρδιά της Ευρώπης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον, καλύτερο δυνατό τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να προωθήσει και τις διεθνείς σχέσεις της. Ε, ε, αυτό είναι το στυλ, αυτό είναι, ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να εργαστούμε μέχρι τον Μάιο του 2015. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την έκθεση αυτή ε, παρά μόνο σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής πρόκλησης. Διότι δεν θέλουμε να περιοριστούμε μόνο στα σύνορα της Ιταλίας, της φιλοξενούσας χώρας, αλλά όσο περνάει ο καιρός θεωρούμε ότι εάν δεν είναι ουσιαστικά ουσιαστικά ευρωπαϊκή έκθεσή μας θα έχει χάσει το στόχο της. Γι' αυτό θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και ε, στηριζόμαστε και στην βοήθειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μαρτίνα και ευχαριστώ και όλη την αντιπροσωπεία της Ιταλικής κυβέρνησης. Ένα λεπτό διάλειμμα, θα ξαναρχίσουμε στις... Ε, 10 για, με, τα, με, τα επόμενα, με το επόμενο θέμα που είναι περιφερειακό σήμα ποιότητας. Ένα λεπτό διάλειμμα. Συνεχίζουμε συνάδελφοι. Σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Περιφερειακό σήμα ποιότητας προς βελτίωση των πρακτικών της αγροτικής οικονομίας. Συναδελφοί, συζητάμε για μια τροπολογία πρωτο, ιδέες πρωτοβουλίες, του συναδέλφου μας ε, κυρίου Ερίκα Ανδριέ. Αυτή η έκθεση παρουσιάζει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ε, περιοχών όπου συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες και το περιφερειακό σήμα ποιότητας ε, πιστεύουμε ότι μπορεί να παίξει ιδιαίτερη σημασία. Ο, το λόγο τον έχει ο Έρικ και μετά θα δούμε ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Έρικ, έχει το λόγο. <clears throat> Euh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή δεν αφορά μόνο ειδικά τη γεωργία και μόνο, αλλά θέτει γενικότερα το θέμα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Διότι οι οικονομικές αλλαγές που σημειώνονται στην Ένωση σημαίνουν ότι πρέπει να μιλήσουμε για κάποιο νέο μοντέλο ανάπτυξης για όλη την Ήπεθρο. Νομίζω ότι η διατήρηση των γεωργών στη δραστηριότητά τους απαιτεί κατ' εμένα να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για εκμετάλλευση προς όφελός τους της παγκοσμιοποίησης. Καταρχήν να λύσω ένα πρόβλημα που μπορεί να δημιούργησε σύγχυση στο αρχικό κείμενο ως προς το σήμα. Ορισμένοι θεωρούν ότι αντιτίθεται η πρόταση αυτή στα σήματα ποιότητας που υπάρχουν ήδη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το ποιοτικό περιφερειακό σήμα θέλει να καλύψει τις προσπάθειες όλων όχι μόνο στην παραγωγή αλλά και στις υπηρεσίες. Όλοι οι τομείς που έχουν σχέση με την ζωή στην Ήπεθρο θα καλύπτονται. Το σήμα λοιπόν αυτό θα καλύπτει όλους τους παράγοντες ιδιωτικούς και δημόσιους για να διασφαλιστεί έτσι μία σφαιρική βιώσιμη ανάπτυξη όλων των περιφερειών με όλους τους τους πόρους και τα υπάρχοντα σήματα επομένως. Δεν υπάρχει θέμα εδώ υποκατάστασης ή ανταγωνισμού, αλλά συνέργειας και συμπληρωματικότητας γύρω από έναν κοινό στόχο. Το διακύβευμα εδώ είναι να φύγουμε από μία ανατομέα αντίληψη που απομονώνει τον κάθε τομέα και να καταλήξουμε σε μια εταιρική σχέση μεταξύ τομέων που να δημιουργεί και περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Είναι νομίζω φανερό ότι η γεωργική δραστηριότητα είναι ουσιώδης για την επιβίωση των περιφερειών αλλά πρέπει να έχει και το κατάλληλο κλίμα και περιβάλλον για να αναπτυχθεί διότι η γεωργία από μόνη της δεν αρκεί για να διατηρηθεί η ζωή της υπαίθρου. Υπάρχουν παραδείγματα που δείχνουν ότι υπάρχουν καινούργια, μπορεί να εφαρμοστούν καινούργια πρότυπα ανάπτυξη στη Γαλλία ας πούμε, στο νότο ιδιαίτερα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας, στην Ισπανία, το Κοντάδο, στη Βάλε Ούμπρα, στην Ιταλία. Υπάρχουν τα παραδείγματα και το πιο ολοκληρωμένο παράδειγμα που γνωρίζω είναι των περιοχών των καθαρών που είναι και η περιοχή που γνωρίζω καλύτερα, γιατί από το 80 ασχολούμαι με αυτές. Συνεννοούνται όλοι οι παράγοντες μιας περιφέρειας, εκεί σε τρεις γαλλικούς νομούς, γύρω από έναν κοινό ιστορικό στόχο και σήμερα πάνω από 35 οικονομικές δραστηριότητες συνεργάζονται γύρω από την ε, εφαρμογή αυτού του σήματος το γάλα, το κρασί, το βόλιο κρέας, το χείριο κρέας, τα τυριά, τα κάμπινγκ, τα ξενοδοχεία, όλα. Αλλά και πέρα από αυτά μπορούμε να μιλήσουμε και για τη βιοτεχνία και το εμπόριο και να βρούμε εκεί παράγοντες που να ενδιαφέρονται για αυτό το σήμα ποιότητος. Όλα αυτά βασίζονται σε μια χάρτα με βάση μια εταιρική σχέση γενικότερη και συγκεκριμένους κανονισμούς και χάρτες για συγκεκριμένα προϊόντα. Έτσι γίνεται μια δικτύωση όλων των προϊόντων και παραγωγών και διευκολύνεται και η απασχόληση. Το όφελος δεν είναι μόνο οικονομικό. Επιτρέπει τη διασύνδεση μεταξύ των παραγόντων και τη συνεργασία τους καθώς και την αλληλεγγύη τους. Η βοσκή είναι αλληλέγγυη με τους παραγωγούς, η παραγωγή με τους μεταποιητές και εκείνη με όλη την υπόλοιπη κοινωνική αλυσίδα. Έτσι δημιουργούνται νέοι δεσμοί στην Ήπεθρο. Αν ήθελα να τα πω ως παραβολή θα χρησιμοποιούσα το παράδειγμα του αργαλιού όπου συνδυάζονται τα νήματα όπως οι χασάπιδες με τους μπακάλιδες. Και όσο πιο σφιχτή είναι η κόμπη, τόσο πιο αλληλέγγυη είναι τα διάφορα επαγγέλματα. Δεν μιλάμε για ανταγωνισμό λοιπόν, αλλά για συνέργεια. Και αυτήν τη συνέργεια θεωρούμε, αυτή η συνέργεια δημιουργεί όλα τα ωφέλη. Και εμείς γνωρίσαμε στις περιφέρειές μας την κρίση στο χείριο κρέας η οποία όμως κρίση ήταν μικρότερη στις δικές μας περιφέρειες γιατί υπήρχαν αυτοί οι δεσμοί μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών οι οποίοι ήξεραν ότι πρόκειται για προϊόντα υψηλής ποιότητας και μάλιστα και με ιστορική αξία. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα μεταξύ άλλων που μπορεί να δείξει πόσο ωφέλιμα μπορεί να είναι αυτά τα νέα πρότυπα. Υπάρχουν ήδη ορισμένα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή αυτής της ποιοτικής παραγωγής. Κυρίως η κοινοτική πρωτοβουλία Leader. Εξάλλου θα γνωρίζετε ότι στο εξής μπορεί κανείς να γενικεύσει τέτοιες εμπειρίες στο σύνολο χωρών, σε ολόκληρες χώρες, καθώς και σε αστικές περιοχές έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη χρηματοδότηση και κινητοποίηση πολλαπλών ταμείων. Επίσης μπορούν να εφαρμοστούν θεματικά προγράμματα για να κινητοποιήσουμε περισσότερα ταμεία. Αλλά νομίζω ότι είναι κυρίως ωφέλιμο εδώ στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης να αναγνωριστεί επίσημα η σημασία ενός περιφερειακού σήματος ποιότητας ευρωπαϊκού επίπεδου ώστε <clears throat> τα περιφερειακά προγράμματα να εφαρμόζονται πληρέστερα και να ολοκληρώνεται έτσι η αγορά αγαθών και υπηρεσιών και περιφερειακά. Είναι μια αναγνώριση περιφερειακών προτύπων ανάπτυξης και μάλιστα βιώσιμων που να λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο τη γεωργία αλλά όλη την οικονομική δραστηριότητα όλων των τομέων που δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο. Ξέρω βέβαια, καταλαβαίνω ότι αυτή η έννοια της ανάπτυξης ξεπερνάει τα απλά γεωργικά θέματα. Και γι' αυτό θα ακούσω ό,τι παρατηρήσεις μπορούν να έχουν οι συνάδελφοι για να βελτιωθεί η πρόταση που σας κάνω σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Ερίκο. Και τώρα πρώτα ο Έρικ Ντόφμαν και μετά ο Εράν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι πολλά χρόνια στον τομέα του Λίντερ, όπως είπε και ο συγητής, υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας και πολλά ενδιαφέροντα μοντέλα έχουν αναπτυχθεί και πιστεύω ότι θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο μέλλον αυτή η συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων της γεωργίας και πέραν της γεωργίας. Και όλα αυτά βέβαια δεν μπορεί παρά να είναι θετικά. Στην μεταρρύθμιση της, ε, του δεύτερου πυλώνα της ε, ΚΓΠ ήδη αναφέρονται αυτά, δεν πρόκειται να ξαναεφεύρουμε τον τροχό. Τώρα υπάρχει αυτή η πρόταση για τις νέες περιφερειακές αγορές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε ένα σύστημα σημάτων ποιότητας που έχει διάφορες διαστάσεις. Προστατεύουμε γεωγραφικά στοιχεία, την προέλευση, ότι είναι ορεινή ε, μια παραγωγή, ένα προϊόν και στο παρελθόν και η Κομισιόν ε, έκανε μεγάλες προσπάθειες όλες αυτές τις ιδέες για διάφορα σήματα που πλανώνται και που δεν βασίζονται σε ε, ενδείξεις ποιότητας να τις αποκλείσει, να απλουστεύσει την κατάσταση. Πριν από μερικούς μήνες, μάλλον έχει περάσει χρόνος από τότε, συζητήσαμε στην Επιτροπή μας την μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για αυτά τα, σήμα ποιότητα, τα σήματα ποιότητας και είχαμε τότε διαπιστώσει πόσο λίγα καταλαβαίνει ο καταναλωτής από τις ήδη υπάρχουσες, από τα ήδη υπάρχοντα σήματα. Τώρα αν εισαγάγουμε και άλλα σήματα που δεν είναι σαφές ε, τι ποιότητα καταδεικνύουν. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Η ιδέα είναι να λέμε ότι ένα προϊόν παράγεται από κάποια περιοχή χωρίς να έχει καμία σχέση με την ποιότητά του. Με αυτόν τον τρόπο θα προκαλέσουμε πλήρη σύγχυση στον καταναλωτή, δεν θα καταλαβαίνει πλέον ουδέν. Ήδη στα, στα πλαίσια του δευτέρου πυλώνα μπορούμε να αναφερθούμε με κάποιες προϋποθέσεις στην προέλευση, τη γεωγραφική ενός προϊόντος. Ειλικρινά δεν έχω την εντύπωση ότι αυτά τα προτινόμενα για νέα σήματα ποιότητας, προέλευσης κτλ. θα πρέπει να επεκταθούν περισσότερο. Δεν νομίζω ότι έτσι πραγματικά εξυπηρετούμε τον καταναλωτή, ότι θα καταλαβαίνει περισσότερα δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνει σήμερα και πραγματικά δεν θα ήθελα μια που τώρα έχουμε ήδη συγκεκριμένα σήματα προστατευόμενης, προέλευση κτλ. να υπάρξει για αυτούς που έχουν ήδη κατοχυρώσει αυτά τα σήματα νέος ανταγωνισμός. Γιατί αυτό θα αποδυναμώσει την σημασία των υπαρχόντων σημάτων. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι έχει έννοια, τι πραγματικά βοηθάει τις επιχειρήσεις, τι βοηθάει και τι θίγει αυτούς που ήδη μπορεί να είναι πολύ επιτυχημένοι. Έχουμε ε, προστατεύσει την γεωγραφική προέλευση ήδη, η γεωγραφική ένδειξη, δεν θα πρέπει να τα αποδυναμώσουμε όλα αυτά. Δεν εξυπηρετούμε έτσι την ευρωπαϊκή γεωργία. Ωραία, ευχαριστώ. Έμπερτ, Άντερ Γκαρσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμμερίζομαι την άποψη του συναδέλφου μου, Herbert Ντόρτμαν, για την υπόθεση αυτή, κύριε Άντριο. Λέτε εσείς από την αρχή ότι δεν έχετε καμία πρόθεση μέσω αυτής της έκθεσης πρωτοβουλία να αποδυναμώσετε τις ε, προστατευόμενες ε, ε, προελεύσεις και τα λοιπά, αλλά στο σημείο 7 της έκθεσής σας εσείς λέτε ότι καλούμε την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη γεωγραφική προέλευση που να βασίζεται σε αντικειμενική ε, αποτίμηση της ε, ε, γεωγραφικής διακυβέρνησης και διαχείρισης. Έχουμε ήδη αυτές τις παραδοσιακές ενδείξεις. Εάν λοιπόν μιλάμε μόνο για αγροδιατροφικά προϊόντα, έχουμε ήδη τα καλύτερα όργανα στη θέση μας και λειτουργούν. Έχουμε την ονομασία προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Είναι αυτές οι δύο μάρκες, αυτά τα δύο σήματα ποιότητας, που λειτουργούν πολύ καλά από όλη μας την κοινή γεωργική πολιτική. Σε, αυτήν, αυτές βασίζονται οι ε, παραγωγοί για να μπορέσουν να διαθέσουν τα προϊόντα τους εντός και εκτός της Ένωσης. Γι' αυτό σας παρακαλώ να βελτιώσουμε αυτά τα εργαλεία που ήδη έχουμε, που ήδη λειτουργούν, αυτά τα δύο που ανέφερα, αλλά σε καμία περίπτωση να μην προσθέσουμε και άλλες πληροφορίες και άλλα λογότυπα και άλλες διοικητικές διαδικασίες και παγίδες. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνουμε αυτά που έχουμε. Να καταργήσουμε βέβαια υπερβολική γραφειοκρατία, αλλά να μην προσθέσουμε προβλήματα. Επιπλέον λέτε ότι δεν θα προκαλέσει σύγχυση. Εγώ νομίζω ότι θα προκαλέσει. Γιατί έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή μας ακριβώς όταν συζητήσαμε τα θέματα ποιότητα το πακέτο μέτρων για την ποιότητα, ήταν ακριβώ ότι υπήρχε ήδη υπερβολική νομοθεσία, υπερβολικά μέσα, που ήδη δεν τα καταλαβαίνουν οι καταναλωτές. Αφού ήδη έχουμε πολλά και αφού δεν λειτουργούν καλά και δεν έχουμε καλή διαχείριση της πληροφόρησης που ήδη υπάρχει για να λαμβάνει ο καταναλωτής την πληροφόρηση, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν ειδήρια ετικέτες για περιφερειακή προέλευση. Τι συζητάμε τώρα. Να αναφέρουμε πού προέρχεται. Μα υπάρχει, υπάρχει. Όλες οι περιφέρειες έχουν δυνατότητα να αναγράψουν ότι ένα προϊόντο έρχεται από τις Αζόρες, όπως μιλάγαμε προηγουμένως, ή από τη Ριόχα, ή από τον Μπορντό, ή από το Άλτο Άντιτζε. Όλοι μπορούν να το πούν ήδη, να το αναφέρουν. Θα μπορούσαμε ίσως να απαιτήσουμε μια σειρά από συγκεκριμένα ε, στοιχεία σε αυτές τις ε, περιφερειακές ετικέτες. Αλλά τώρα ε, δεν ξέρω να συζητάμε μόνο για αγροτροφημικά προϊόντα ή συζητάμε για κάτι ευρύτερο ε, τότε θα έπρεπε να το συζητήσει η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να αναλάβουμε εμείς ως άγκρη πρωτοβουλία. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να περιοριστούμε, να ζητήσουμε ενδεχομένως πιο αυστηρή αναγραφή, πιο απαιτητική, αλλά να μην ε, εισαγάγουμε και άλλα στοιχεία, γιατί αρκεί η πληροφόρηση που ήδη μπορεί να αναφερθεί. Ευχαριστώ πολύ. Πατράου Νέβες και μετά η Ευχαριστώ. Εγώ υποστηρίζω θερμά τις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. Είμαι πεπισμένη ότι μια τέτοια ολοκληρωμένη παρέμβαση μπορούν να βοηθήσουν την ε, καλύτερη χρήση των πόρων και του ανθρωπίνου δυναμικού και να οδηγήσουν σε περισσότερη αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, λοιπόν, το θέμα που συζητάμε αυτή τη στιγμή μου δημιουργεί μεγάλες και σοβαρές αμφιβολίες για το εάν και κατά πόσο η παρέμβαση που προτείνει ο εισηγητής είναι η καλύτερη μορφή αντιμετώπισης του θέματος αυτού. Καταλαβαίνω βέβαια ότι ο εισηγητής έχει διαπιστώσει τα προβλήματα που έχουν αναφέρει και άλλοι συνάδελφοι. Και εγώ θα τα αναφέρω. Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο εισηγητής ξέρει ότι μπορεί να προκληθούν κάποιες ε, επικαλύψεις, κάποιες συγχύσεις, κάποιες συγκρούσεις. Οπότε, προσπαθεί να παρακάμψει τα προβλήματα στην ουσία. Οπότε δεν με πείθει. Γιατί ε, αν συζητάμε για ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων, σε αυτή την περίπτωση η τομεακή προσέγγιση νομίζω ότι είναι η μόνη που ε, μπορεί να μας χορηγήσει αρκετές εγγυήσεις για να ε, δώσουμε σωστή πληροφόρηση στο καταναλωτή. Σοβαρή πληροφόρηση. Λοιπόν, τι εννοούμε σοβαρή. Εάν μία ετικέτα καλύπτει υπερβολικά ευρύ πεδίο πληροφόρησης, τότε δεν θα δώσει πολύ ουσιαστική πληροφόρηση. Οπότε, από τη μία αυτό θα θίξει τα προϊόντα που είναι πραγματικά υψηλής ποιότητας, και που σε κοινοτικό επίπεδο ήδη έχουν δυνατότητες να αναφέρουν με τρόπο που να περνάει στο καταναλωτή ε, την ποιότητά τους ενώ τα άλλα προϊόντα που δεν είναι τόσο υψηλής ποιότητας τα άλλα λοιπόν προϊόντα θα επωφεληθούν από αυτήν την ε, γενική εντύπωση ποιότητας που θα ε, συνδεθεί με κάποιο σήμα χωρίς την ουσία να παρέχουν αυτή την ε, ποιότητα. Έτσι δεν εγγυόμεθα την ποιότητα. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος να απογοητεύσουμε τους παραγωγούς διότι αυτοί που, θα, αυτοί που παράγουν πραγματικά ε, ε, ποιοτικά προϊόντα θα θεωρήσουν ότι αδικούνται. Ξέρετε, οι καταναλωτές στην εποχή μας κατακλείζονται από κάθε είδους ε, σήματα, λογότυπα, ενδείξεις. Άλλο ένα να δημιουργήσουμε. Δεν είμαι πεισμένη. Νομίζω ότι τα υπερβολικά σήματα θα σκοτώσουν τελικά τα σήματα. Πρέπει, πιστεύω, να περιορίσουμε τον αριθμό σημάτων και ενδείξεων για να έχουν αξιοπιστία αυτά τα οποία αναφέρονται. Έχουμε ήδη τις ε, προστατευμένες και ελεγχόμενες ονομασίες προέλευσης, ε, τις ενδείξεις γεωγραφικής, ε, και ποιο... γεωγραφικής προέλευσης και ποιότητας. Εάν βάλουμε και άλλα, στην ουσία τα αποδυναμώνουμε όλα αυτά. Δεν έχω την εντύπωση ότι θα προσφέραμε τίποτα περισσότερο μέσω αυτής της οδού. Ξέρω βέβαια ότι ο εισηγητής έχει συνέστηση των δυσχεριών που θα μπορούσαν να προκύψουν. Θα τον παρακαλούσα λοιπόν να λάβει υπόψη παρακαλώ τα σχόλιά μας γιατί ξέρετε βεβαίως όλοι έχουμε κοινό στόχο να προωθήσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε και επί της ουσίας. Άγνιου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς Ευχαριστώ τον συγητή, τον σύντροφο Ερικ για την εργασία που περιέχεται στην έκθεσή του. Νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε την άποψη ότι χρειάζεται να έχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα στον τομέα της υπαίθρου, να έχουμε κοινέ ενέργειες στον οικονομικό, τον κοινωνικό και άλλους τομείς για να αναπτύξουμε την Ήπεθρο να ε, αναπτύξουμε τη γεωργία από όλε τι απόψεις. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τα προγράμματά μας. Οτιδήποτε βοηθάει αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό είναι ελκυστικό. Όπως το αναφέρει και η έκθεση να συμπεριληφθεί ο τουρισμός, ε, η στήριξη στις γεωργικές δραστηριότητες, την ε, οικογενειακή γεωργία κτλ. Στις οικογενειακές δραστηριότητες. Όπως όμως είπαν και οι προηγούμενοι, θα αναφερθώ σε, αυτή τη σήμα, σε αυτό το σήμα. Πριν από ένα χρόνο ολοκληρώσαμε μία έντονη συζήτηση για τα συστήματα ποιότητας, για τα θέματα που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας. Ήμουν μάλιστα εγώ, είχα την τιμή να είμαι εισηγήτρια. Σε όλη αυτή τη συζήτηση κάναμε ανταλλαγή απόψεων, ανησυχιών, και μία από τις κύριες ανησυχίες που αναφέρθηκε από πολλούς ήταν ακριβώς ε, αυτή η πολυπληθής, ε, αυτή, ε, αυτές οι όλο και περισσότερες μάρκες και σήματα που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στον καταναλωτή. Μετά την αναθεώρηση της οδηγίας για το θέμα αυτό και την εφαρμογή της νέας οδηγίας για τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας, είναι σαφή η κατάσταση και οργανώσεις παραγωγών και όλοι αυτοί που αξιοποιούν αυτά τα σήματα έχουν μια σαφή αντίληψη για το ποιε είναι οι αυστηρές προδιαγραφέ ποιότητας τις οποίες πρέπει να συμμορφούνται. Και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής πληροφόρηση του καταναλωτή προσπαθούμε να γνωρίζει τι προσθεμένη αξία έχουν τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτά τα συστήματα ποιότητα, γεωγραφικέ ενδείξει, προστατευόμενε κτλ. Ούτω ώστε οι καταναλωτέ να καταλαβαίνουν τη διαφορά μεταξύ αυτού του συστήματο και άλλων συστημάτων ποιότητα που δεν είναι τόσο αυστηρά και που δεν πληρούν τις ίδιε προδιαγραφές. Αυτή η ανησυχία μας ε, αναφέρθηκε και σε συναντήσεις που κάναμε με παραγωγούς σε διάφορες χώρες. Γιατί σήμερα Αυτά τα σήματα περιφερειακής ποιότητας υπάρχουν. Έχουν γίνει όλο και περισσότερα. Έχουν πολλαπλασιαστεί σε διάφορες περιφέρειες και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ένα σήμα ποιότητας που δεν σημαίνει στην ουσία ότι πληρούνται οι αναγκαίες προδιαγραφές. Οπότε αισθάνονται απροστάτευτοι οι παραγωγοί που τηρούν αυτές τις προδιαγραφές και προκαλείται και σύγχυση στον καταναλωτή. Όταν πάει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει τόσα λογότυπα, τόσες μάρκες, τόσα σήματα. Οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση. Στην έκθεση αυτή να εμβαθύνουμε τις προτάσεις ολοκληρωμένων προτάσεων τις ολοκληρωμένες προτάσεις για ανάπτυξη της υπαίθρου με ένα αυστηρό σύστημα ποιότητας και η παραγωγή που πληρούν τις θετικές αυτές προδιαγραφές που προσθέτουν προστιθέμενη αξία, που προσθέτουν αξία, θα πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στην πληροφόρηση του καταναλωτή. Αυτό σημαίνει να αναφέρεται σαφώς ποιό συμμετέχει στα συστήματα ποιότητας. Ελπίζω λοιπόν ότι μέσω της υποβολής τροπολογιών θα δούμε πώς θα τροποποιήσουμε αυτήν την ε, έκθεση. Ξαναλέω, υποστηρίζω πλήρως τους παραγωγούς που συμμορφούνται με προδιαγραφές για ε, συγκεκριμένα σήματα και να συνδυάσουμε αυτή την προσπάθεια με τις στρατηγικές μας εντός του Leader για την ανάπτυξη πέτρου ή άλλες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Ράτσε. Τώρα ο Άγνιο και μετά Γιώχανσον. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα αυτό του περιφερειακού σήματος ποιότητας είναι πολύπλοκο και μπορεί να περιέχει πολλές παγίδες. Θα σας δώσω τρία παραδείγματα που μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση. Μερικές φορές υπάρχει ε, μια γενική, ένα γενικό προϊόν όπως το τυρί Τσέσερ που είναι από την κομιτεία του Τσέσερ αλλά πρόκειται στην ουσία για τον τρόπο παρασκευής του τυριού. Δεν είναι ανάγκη να προέρχεται από το Τσέσαρ. Το όνομά του δείχνει μια, έναν τρόπο παραγωγής. Υπάρχουν όμως και πιο συγκεκριμένα σήματα και είδη τροφίμων που μπορεί να έχουν πιο μεγάλη, πιο μεγάλη σχέση με τον τόπο παραγωγής. Τότε πρέπει να έχουν την άδεια της Ένωσης και τον έλεγχο μήπως καμία άλλη ενωσιακή χώρα έχει αντιρρήσεις. Εγώ δεν αφωνώ με αυτό. Πρέπει η χώρα να αποφασίζει. Έπειτα. Η περίπτωση όπου είναι πολύ σημαντική ιστορική γεωγραφική προέλευση όπως ας πούμε πατάτες Φιλανδίας που οφείλονται, η ποιότητά τους οφείλεται στην ποιότητα του εδάφους ας πούμε έχουν μαύρο έδαφος εκεί. Όσο διαφορετικές και να είναι οι πατάτες έχουν την ίδια εμφάνιση. Τέλος Υπάρχει το θέμα του τόστ που λέγεται Wells Rarebit. Αυτά είναι όλα θέματα της κάθε χώρας και δεν πρέπει να παρεμβαίνει η μία στις παραδόσεις της άλλης. Ευχαριστούμε Άγνιο, Γιώχανσον και μετά Κλάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν νομίζω ότι είναι πολύ θετικό ότι στην έκθεση αυτή μπορούμε να προβλέψουμε συνεργασία, περιφερειακή συνεργασία και μεταξύ χωρών. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για τη Γεωργία αυτό. Διότι πρέπει οι αγροτικές περιφέρειες να μην υποστούν ζημίες λόγω έλλειψης περιφερειακής συνεργασίας. Ευχαριστώ λοιπόν τον συγκητή για όσα έχει κάνει και συγχαίρω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ασχολείται με αυτό το θέμα. Τώρα, συγκεκριμένα για την ποιότητα και το σήμα αυτό ποιότητος. Έχω μερικά σχόλια και απορίες να σας εκφράσω θα χρειαστεί και ενούργια άλλη συζήτηση όταν εξετάσουμε τις τροπολογίες βέβαια. Η συνεργασία μεταξύ κύριου εισηγητή και σκιωτών θα μας δώσει αυτή την ευκαιρία. Όπως και άλλοι συνάδελφοι θα ήθελα και εγώ να μιλήσω τώρα για αυτό το σήμα ποιότητος. Είναι κάτι, μια έννοια που είναι γενικά αποδεκτή ή κάτι καινούριο. Στο σημείο 7 λέει ότι η Κομισιόν πρέπει να καθορίσει την έννοια αυτή του Ευρωπαϊκού Σήματος Ποιότητος. Ε, όπως και οι άλλοι λοιπόν, αναρωτιέμαι και εγώ, τι άλλες έννοιες συγκρίσιμες υπάρχουν πέρα από αυτήν την, αυτό το Ευρωπαϊκό Σήμα Περιφερειακής Ποιότητας, Περιφερειακό Σήμα Ποιότητας. Γίνεται λόγος επίσης για αγροτικά προϊόντα, για υπηρεσίες, για τον τουρισμό. Αφού λοιπόν μιλάμε για περιφερειακό σήμα ποιότητας, θα έπρεπε να πούμε ότι είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται περισσότερη περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. και εθνικά και περιφερειακά μπορούν να βρεθούν τρόποι ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας είναι και αυτό σημαντικό και θα γίνεται όλο και σημαντικότερο στις νέες δημοσιονομικές περιόδους. Τώρα ένα θέμα αρχής που θέτει ο ίδιος ο εισηγητής πρέπει όχι να χρησιμοποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία που έχουμε για την ανάπτυξη της υπαίθρου ή μήπω χρειαζόμαστε καινούρια όπως λέει ο εισηγητής. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε, να το ξανασυζητήσουμε. Γενικά λοιπόν το σχόλιο μου είναι ότι είναι πολύ θετικό όπως λέει και ο εισηγητής να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία σε οριζοντίως σε περιφερειακό επίπεδο και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες που έχουμε. Δεν είναι θέμα απλώς οικονομικό, αλλά και η κοινωνία των πολιτών ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της υπαίθρου ή την ανάπτυξη στην υπαίθρου. Θα επανέλθω όμως όπως είπα στις επόμενες συζητήσεις μας όταν θα μιλήσουμε για τις τροπολογίες. Και αυτή η παράγραφος που ανέφερα, η 7, για το προτινόμενο νέο σύστημα και την επίσημη αναγνώριση του σήματος είναι η πιο ενδιαφέρουσα. Αυτό ίσως θα συζητήσουν οι τροπολογίες, θα δούμε. Η κυρία Κλάς, ευχαριστώ. Οι εκθέσεις πρωτοβουλίας δεν έχουν νομοθετική επίπτωση, αλλά ε, scripta Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε, όπως και οι άλλοι προηγούμενοι, ε, κριτικά το κείμενο αυτό και συμφωνώ με όλους όσους ε, εξέφρασαν κάποιους φόβους και να είμαι σαφής. Δεν χρειαζόμαστε, αυτό ακριβώς που δεν χρειαζόμαστε είναι και άλλο σήμα ποιότητας. Και δεν μπορούμε ούτε καν να κάνουμε να λειτουργήσουν σωστά και να γίνουν γνωστά αυτά. Οι καλές προθέσεις δεν επαρκούν πάντα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε. Μήπως με αυτήν την έκθεση ε, κάνουμε λάθος και, και ε, δημιουργήσουμε πράγματα τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Γιατί τα πράγματα ε, ήδη πηγαίνουν καλά. Βέβαια, ε, έχει καλές προθέσεις, είναι σαφές ο εισηγητής. Πρέπει όμως να βρούμε έναν τρόπο, ούτω ώστε αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας να διαμορφωθεί έτσι, ούτω ώστε αυτά που ήδη έχουμε να συνεχίσουν να εφαρμόζονται σωστά γιατί νομίζω ότι οι εκλογείς μας δεν θα ενθουσιαστούν και τόσο πολύ εάν με βάση την παράγραφο 7 απαιτήσουμε έναν κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, προέρχομαι από μια περιοχή που έχει έντονη γεωργική δραστηριότητα. Από μια περιοχή η οποία καταλαβαίνει καλά τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα εφαρμόζει. Και υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες ήδη. Υπάρχουν και για το Μοζέλα και για την περιοχή του Άιφελ και δεν αφορά μόνο τη γεωργία, όχι μόνο τη βιομηχανία, όχι μόνο τον τουρισμό, όχι μόνο τον πολιτισμό. Όλοι αυτοί οι τομείς συνεργάζονται σε αυτή την περιοχή για να υπάρχει αυτή η μάρκα Μοζέλα, η μάρκα Άιφελ ασχολούνται, η πολιτικοί με αυτό, οι... αυτοί που εργάζονται στη γεωργία, στον τουρισμό κτλ. Σας παρακαλώ. Όχι άλλοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Πώς θα τους πείσουμε ε, στις περιοχές μας να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ, όχι την παράγραφο 7 όπως είναι τώρα. Να αναφέρουμε πρακτικά παραδείγματα, πώς μπορούμε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας πώς μπορούμε να διευρύνουμε σε περιφερειακό επίπεδο την προσπάθεια αυτή και να την ενισχύσουμε. Δεν θα καθορίσουμε εδώ ότι είναι περιφέρεια. Παρακαλώ, αυτό θα ήταν αντίθετο στο στόχο μας. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας παρακαλώ να ξανασκεφτούμε τι θέλουμε να περιέχει αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας να μην ε, εφαρμόσουμε στην Ευρώπη ένα στενό κορσέ που δεν θα τη επιτρέπει πια να αναπνεύσει. Αυτό θα καταστρέψει τα πάντα αντί να ε, βελτιώσει την κατάσταση και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κλάς για την, ε, με την παρέμβαση αυτή. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών από την Επιτροπή μας. Θα ήθελα να ρωτήσω η Κομισιόν, έχει να πει τίποτα, ο κύριος Μισελ Εράτη είναι παρόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Επιτροπής ήθελα να υπογραμμίσω ότι με το σύστημα προστασίας γεωγραφικών ε, προελεύσεων και ποιότητας ήδη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σήματα και διαδικασίες για να υποστηρίξουν, ε, υποστηρίξουμε προϊόντα τα οποία έχουν χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας. Μόνο η ε, οι ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης και ποιότητας έχουν το δικαίωμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναφέρονται σε αυτή την περιφερειακή εξειδίκευση. Για τα θέματα, τα συστήματα ποιότητας που δεν συνδέονται με την προέλευση, δηλαδή που είναι ανοιχτά για το σύνολο των προϊόντων, το άρθρο 17 του μελλοντικού κανονισμού για την ανάπτυξη της υπαίθρου που υιοθετήθηκε θα προβλέπει μια δυνατότητα αναγνώρισης για συστήματα ποιότητας τα οποία θα υιοθετούν ε, τα κράτη-μέλη. Μία προϋπόθεση για την υποστήριξη είναι ότι το σύστημα να μην περιορίζεται μόνο στα προϊόντα μίας περιοχής αλλά να είναι ανοιχτό στο σύνολο των προϊόντων. Εν τέλει, η Κομισιόν έχει υιοθετήσει και, μία, και κατευθυντήριες γραμμές για τα σήματα ποιότητας και τα περιφερειακά σήματα ε, από το 2010 με, ε, και υπάρχει σύστημα ε, εθελούσιας πιστοποίησης για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα. Έχουμε δηλαδή ήδη μία ανακοίνωση που αφορά το θέμα αυτό. Η δημιουργία μιας, ενός περιφερειακού, σήμα, ε, περιφερειακού σήματος ποιότητας για το σύνολο των προϊόντων μπορεί να θίξει τις ε, Ενδείξει ε, και τις ονομασίες γεωγραφικής προέλευση στις συγκεκριμένε περιοχές. Μια τέτοια, ένα τέτοιο σήμα μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση των καταναλωτή. το σήμα της, ε, του περιφερειακού σήματο Ποιότητα στην Ευρώπη θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θίγει και, την, ε, και το άρθρο 34 μάλλον κατά πόσον θίγει την Ευρωπαϊκή Νομολογία με βάση το άρθρο 34 του κανονισμού για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ενθουσιώδης με την, σημασία, με την δημιουργία του Περιφερειακού Σήματος Ποιότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κομισιό, τον κύριο Εράτα και ο Ερίκ Αντρέ, αν έχει το λόγο. Ερίκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των, συναδέλφων που πήραν το λόγο, διότι ο καθένας κατάλαβε εδώ ότι το θέμα μας δεν είναι το σήμα, δεν είναι το σήμα το οποίο ήθελα να υπογραμμίσω, αλλά η ανάπτυξη της υπαίθρου. Μιλήσαμε για γεωργικά σήματα, δεν είναι αυτό το, θέμα μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε όλα τα σήματα προστασίας της ποιότητας που θέλουμε. Αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να διατηρήσει την ε, δραστηριότητα στο σύνολο το, της περιφέρειάς μας, των περιοχών μας. Είναι πιο περίπλοκο το θέμα και όπως είπαν πολλοί ομιλητές πρέπει να βρούμε μεθόδους έτσι ώστε όλοι ε, οι οποίοι ασχολούνται ε, και απασχολούνται στον τομέα αυτό να καταλάβουν την ανάγκη της συνεργασίας. Η γεωργική δραστηριότητα είναι σημαντική, αλλά υπάρχουν και υπηρεσίες, υπάρχουν, ε, υπάρχει τουρισμός, ε, υπάρχει πολιτισμός. Ε, όλοι αυτοί οι κλάδοι, όλοι αυτοί οι τομείς πρέπει να συνεργαστούν. Ίσως να μην εκφράστηκα πάρα πολύ καλά προηγουμένω και το μόνο που να βρήκα είναι το περιφερειακό σήμα ποιότητα. Όμω δεν είναι αυτό το δεν είναι αυτή η καρδιά της έκθεσης, δεν είναι η ουσία της έκθεσης. Ίσως να, βρούμε μια άλλη, να πρέπει να βρούμε μια έκφραση εάν υπάρχει σύγχυση, αλλά δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε το προϊόν και την διαδικασία κτλ. Απλώς θέλω να βρούμε μια μέθοδο έτσι ώστε ο καθένας που λειτουργεί σε, ένα, σε μια περιφέρεια, σε μια περιοχή να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της περιοχής και υπάρχουν περιφερειακά σήματα ποιότητα τα οποία γεννιόνται θέλουμε ή όχι σε όλη την Ευρώπη με οποιονδήποτε τρόπο όπως θέλει ο καθένας και αυτό είναι ει βάρο της ε, ποιότητα, αν θέλετε ε, ε, και των γεωγραφικών προελεύσεων γι' αυτό εμείς πρέπει να προβλέψουμε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε από κοινού να βάλουμε με ένα πλαίσιο και μία μέθοδο έτσι ώστε το περιβάλλον σε αυτές τις δυναμικές που δημιουργούνται ε, σε όλη την Ευρώπη να μπορεί να ελεγχθεί έτσι ώστε να μην έχουμε σύγκριση με τις ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης και ποιότητας. Πρόεδρε, πιστεύω ότι το πρόβλημα πρέπει να τεθεί με διαφορετικούς όρους ε, και όχι έτσι όπως ετέθη σήμερα από τους διαφόρους συναδέλφους ε, ενδεχόμενα, όμως πρέπει, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει στην Επιτροπή Γεωργίας και Γεωργικής Ανάπτυξης. Μιλάμε για τη γεωργία προφανώς και είμαστε τώρα στα τελευταία στάδια της γεωργικής μεταρρύθμισης, όμως θα πρέπει να σκεφτούμε και την ανάπτυξη της υπαίθρου γενικότερα. Όταν σήμερα η ανάπτυξη, η, ο διαχωρισμός ανάπτυξα στην γεωργία και στην ε, ε, γεωργική πολιτική και στην, ε, συγγνώμη, στην ανάπτυξη της υπαίθρου συνδέονται, πρέπει και εμείς να ασχοληθούμε με τον, με χώρο της υπαίθρου, διότι η υπαίθρος οικονομικά και, και αγροτικά είναι ένα σύνολο. Άρα θα πρέπει να βρούμε κάποιες μεθόδους έτσι ώστε να κινητοποιήσουμε, να προκαλέσουμε μια συνεργασία όλων των παραγόντων, όλων των όσων ασχολούνται με τον τομέα αυτό και να, για να έχουν ένα κοινό μοντέλο. Βέβαια είπαμε ότι είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας και ήθελα ακριβώς να κάνω αυτές τις προτάσεις για να ξεκινήσει μια κάποια σκέψη και ε, άκουσα και τον ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ξέρω ότι υπάρχουν τέτοιου είδους ε, σήματα. Εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω έναν ανταγωνισμό, απλώς θέλω να πω ότι πρέπει να σκεφτούμε από κοινού και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έτσι ώστε να ασχοληθούμε περισσότερο με τα θέματα της υπαίθρου και σε αυτή την αντιπαράθεση αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου να ασχοληθούμε με την υπαίθρο. Ευχαριστώ Ερικ, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε και να ε, ακούσουμε ποιες, πώς θα εξελιχθούν όλες αυτές οι ευαισθησίες ε, που ακούστηκαν σήμερα εδώ. Πάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης Σημείο 11. Έλεγχοι και δραστηριότητε που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Συντάκτρια η κυρία Μπρίτα Ρέιμερ. Α, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό Μπρίτα. Μισό. Μου υπενθυμίζει η γραμματεία ότι δεν αναφέρθηκα για την στην προθεσμία κατάθεσης ε, τροπολογιών για την έκθεση του, του ΕΡΙΚ. 1η Οκτωβρίου, 1η Οκτωβρίου η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών, διότι μέχρι τις 25 Νοεμβρίου πρέπει να υποβάλουμε την ε, έκθεση. Λοιπόν, μετά από αυτή την παρένθεση, επανέρχομαι στην ε, έκθεση της Μπρίτα. Ακούσαμε και χτες στην Επιτροπή μας διάφορα θέματα για αυτό το πακέτο τρόφιμα και ζωοτροφές. Είναι ε, ε περίπλοκο το θέμα, γι' αυτό χωρίς ε, ε, καμία καθυστέρηση δίνω το λόγο κατευθείαν στην Μπρίτα. Ξέρετε ότι με, το, με την Επιτροπή Περιβάλλοντος αυτό το θέμα υπάρχει μια αντιπαράθεση και ελπίζω ότι θα τελικά θα καταφέρουμε να έχουμε μία συνάντηση με τον Ματίας Γκρότου, τον πρόεδρο της Επιτροπής, έτσι ώστε να είναι θετικές οι εξελίξεις και τις δύο επιτροπές μας. Ούτως ή άλλως το λόγο να είσαι συμπρίτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα. την έκθεση για αυτούς τους επισήμους ελέγχους. Στόχος της Κομισιόν είναι να εφαρμοστεί καλύτερα ε, να εφαρμοστούν καλύτερα οι κανόνες για την ασφάλεια και την ε, ποιότητα των ε, τροφίμων καθ' όλη τη διάρκεια της αλυσίδας παραγωγής. Θέλει να απλουστεύσει τη διαδικασία και θα ήθελε 70 νομοθετήματα, νομοθετήματα να περιοριστούν σε 5 Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ευρία επίπτωση, πόσο μεγάλο είναι αυτό το πακέτο. Η Επιτροπή θα ήθελε να μειώσει τη γραφειοκρατία και για τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, τις επιχειρήσεις και θεωρεί ότι μειώνοντας την με βάση ε, προδιαγραφές ε, ε, που έχουν εκπονήσει οι επιστήμονες για την, με βάση την εκτίμηση του κινδύνου θεωρεί λοιπόν ότι είναι δυνατόν αυτό με αυτό τον τρόπο θα καταπολεμήσουμε και όλα τα παράσιτα που αντιμετωπίζουν τα φυτά και τα ζώα. Θα βελτιώσουμε λοιπόν τους ελέγχους μέσω της ενίσχυσης των υπηρεσιών των κρατών μελών για να μπορούν να τηρούν τους κανόνες μέσω ελέγχων και τεστ θα ληφθούν μέτρα πιο αποτελεσματικής ε, εφαρμογής και ενημέρωσης ε, των ε, καταναλωτών και των παραγωγών για, τις, ε, για τους κινδύνους. Και θέλουμε να βελτιώσουμε όλη την αλυσίδα. Πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε για τις μικρές επιχειρήσεις, για τις μικρότερες. Είναι πάντα ο κίνδυνος ότι θα είναι υπερβολικό το άχθος για αυτούς. Αυτές θα τις εξαιρέσουμε για να εγγυηθούμε την ανταγωνιστικότητά τους. Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή όλων των ελέγχων κατά των απατών και τα κράτη-μέλη μπορεί να αντιμετωπίσουν και αποτρεπτικά πρόστιμα αν τα συστήματα απατών, αντιμετώπιση των απατών δεν λειτουργούν. Όπως για παράδειγμα ε, το πρόβλημα που είχαμε με το αλογίσιο κρέας. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε μια σειρά από κατεξοδότηση πράξεων. Όταν συνοψίζει κανείς τα 70 σε 5 υπάρχουν ανάγκες τέτοιων κατεξοδότηση πράξεων και πρέπει να δώσουμε ε, εξοδότηση στην Κομισιόν για να κάνει τέτοιες ε, να εκδίδει τέτοιε κατεξοδότηση πράξεις αλλά όταν τι χορηγούμε τέτοιε αρμοδιότητε θα πρέπει να προσέξουμε πού τι χορηγούμε και όταν κάνουν έλεγχο τα κράτη-μέλη πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει συνολικός ε, έλεγχος αυτής της διαδικασίας όχι μόνο από την Κομισιόν, αλλά και με συμμετοχή υποπτική του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να συζητήσουμε και το ύψος ε, των, ε, του κόστους αυτών των προσπαθειών. Βεβαίως, επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την επικουρικότητα. Να εξετάσουμε, λοιπόν, εάν και κατά πόσο είναι αποδεκτή ή είναι δυνατόν να, τα κράτη-μέλη να φέρουν το κόστος αυτών των συμπληρωματικών ελέγχων, να δούμε τι θα πρέπει να τους επιβάλλουμε και τι θα πρέπει να τους επιβάλλουμε. Και σε ορισμένε περιοχέ, σε ορισμένα κράτη που έχουν ομοσπονδιακή δομή, θα πρέπει να κατέβουμε και σε επίπεδο ομόσπονδου κράτου. Είναι πολύ ευρεία λοιπόν η προσπάθεια αυτή. Αυτό είναι καλό αλλά για την ποιότητα και την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων πάντα μας ενδιέφερε όλη η αλυσίδα από τους παραγωγούς μέχρι τους μεταποιητές, τους εμπόρους κτλ. Βέβαια αυτό μπορεί να προκαλέσει ε, περισσότερη αφροκρατία. Να δούμε λοιπόν εάν χρειάζεται να ε, εισαγάγουμε περισσότερες λεπτομέρειες ή απλώς να βελτιώσουμε το υπάρχον σύστημα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να δούμε σε τι βαθμό και με τι τρόπο εφαρμόζεται το υπάρχον δίκαιο στα κράτη-μέλη. Η προσπάθεια απλούστευσης και περιορισμού σε πέντε είναι καλή. Ε, χαίρομαι για το θάρρος της Κομισιόν, αλλά πρέπει να εξετάσουμε αν μπορεί να γίνει αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη και σε τι βαθμό θα μπορούσε αυτό να επηρεάσει ε, νόμους στα κράτη-μέλη που δεν θέλουμε να καταργήσουμε. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Οπωσδήποτε και με τους σκιώδεις συζητητές των πολιτικών ομάδων θα πρέπει να το συζητήσουμε πολύ περισσότερο. Το πακέτο είναι τόσο μακρόπνο που δεν είναι δυνατόν να το αντιμετωπίσουμε πρόχειρα. Θα έπρεπε να υπάρχει τακτική έντονη ανταλλαγή απόψεων γιατί το πακέτο αυτό θα έχει ε, ευρείες επιπτώσεις για τις επόμενες δεκαετίες. Ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσίαση αυτή και ε, προσβλέπω στις ε, παρεμβάσεις και την ε, αρρωγή των συναδέλφων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπρίτα. Η κυρία Γκαρσία ζήτησε το λόγο, δεν βλέπω άλλους. Σημερίζομαι την άποψη της συγγήτρες της κυρίας Άιμερ, να πούμε δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι, καλή αυτή η έκθεση, αλλά περιέχει πολλά στοιχεία Πρέπει να επεκτείνουμε τον τομέα εφαρμογής του κανονισμού σε όλους τους τομείς και σε ορισμένου που είναι εξωτερικοί της διατροφικής αλυσίδας. Παράδειγμα. Οι γεωγραφικές ενδείξεις, οι ενδείξεις ποιότητας είναι ή δεν είναι εντός του πεδίου εφαρμογής. Να το διευκρινίσουμε. Τι σημαίνει επίσημος έλεγχος. Τι σημαίνουν άλλοι επίσημοι έλεγχοι. Γιατί όπως αναφέρατε τώρα δεν είναι σαφές. Εγώ νομίζω ότι αυτό το κεφάλαιο άλλη επίσημη έλεγχη πρέπει απλώς να διαγραφεί. Τελευταία βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια τάση να ε, παράγονται όλο και περισσότερες οι πράξεις και εκτελεστικές πράξεις. Πολύ φιλόδοξη είναι η Κομισιόν. Θέλει να μπλέξει σε τομείς που δεν είναι αρμοδιότητά της και να ε, περιορίσει τις δυνατότητε δράσης άλλων φορέων της Ένωσης όπως το Κοινοβούλιο. Σήμερα στην ε, συζητήση μας, στη συζητήση μας σήμερα είδαμε πως η Κομισιόν μέσω τέτοιων πράξεων προσπαθεί να μας βγάλει από τη μέση. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Ε, με πρόσχημα ότι αυτή είναι πιο αποτελεσματική και πιο ταχύς. Για τους φόρους αυτούς που λένε ότι πρέπει κατευθείαν οι, αρχικές, κατευθείαν οι εθνικές αρχές πρέπει να τους εφαρμόζουν. Ε, στη χώρα μου αυτές οι εθνικές αρχές του Υπουργείου ε, Οικονομίας είναι αρμόδιες για την συλλογή και διανομή συλλογή φόρων και διανομή ε, ενισχύσεων. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να είναι αρμόδια για αυτά τα θέματα. Για τους ελέγχους εξαγωγών. Και αυτή είναι αρμοδιότητα κρατών μελών. Επικουρικότητα. Να... Οπότε η Κομισιόν όταν ζητά αρμοδιότητες και σε αυτό το τομέα υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της με βάση τις συνθήκες. Και τέλος, η Επιτροπή επίσης θέλει να συμμετάσχει και στους ελέγχους που κάνουν τα, οι τρίτες χώρες στις χώρες μέλη πριν ε, εγκρίνουν εξαγωγές. Και εδώ υπερβαίνει τις αρμοδιότητές της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Γκαρσία. Αν δεν ζητάει κανείς άλλο το λόγο, θα δώσω το λόγο στην Κομισιό. Η κυρία Κάρμεν Γκαράου ε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο μόνο σχόλια. Δηλαδή ένα κυρίως ότι η πρόταση αυτή δεν άρχισε, δεν βασίστηκε στο μηδέν, δεν άρχισε από το μηδέν. Υπάρχει ήδη νομοθεσία για επίσημους ελέγχους η 82 του 2004 που ήδη προβλέπει πολλά από αυτά που αναφέρθηκαν από την εισηγήτρια για τις δικαιοδοσίες, για τις αρμόδιες αρχές που θα αναλάβουν τους ελέγχους κλπ. Αυτό είναι το κύριο σχόλιο που ήθελα να κάνω. Τώρα ιδιαίτερα για τις τιμές. Η πρόταση, η νομοθεσία που ισχύει αυτή τη στιγμή επιβάλλει για μερικούς τομείς μόνο αυτούς τους ελέγχους επιπληρωμή. Η πρόταση λοιπόν στοχεύει εδώ να εξισορροπήσει τα πράγματα έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλοι όσοι υποβάλλονται σε έλεγχο και να πληρώνουν τα ίδια δεν προβλέπεται εναρμόνιση του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι τιμές αυτές. Λέει να βασίζεται στο κόστος η τιμή, αλλά επειδή το κόστος είναι διαφορετικό σε κάθε χώρα μέλος, οι τιμές του ελέγχου λοιπόν θα αντικατοπτρίζουν αναγκαστικά το βιωτικό επίπεδο, το κόστος ζωής δηλαδή στην κάθε χώρα μέλος. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα των ε, αναπαραγωγικών υλικών κτλ. Αυτά καλύπτονται ήδη από τον υπάρχοντα κανονισμό. Η μεγαλύτερη αλλαγή που προβλέπει η πρόταση αυτή είναι να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του επίσημου κανονισμού ελέγχων έτσι ώστε όλοι οι έλεγχοι που κάνουν οι αρμόδιες αρχές σε όλη τη διατροφική αλυσίδα και της πρωτογενούς παραγωγής και της μεμπορίας όλοι αυτοί οι τομείς να διέπονται από τους ίδιους κανόνες για τους επίσημους ελέγχους που θα κάνουν οι χώρες μέλη. Όσο για τις κατεξουσιοδότηση πράξη. υπάρχει εδώ μια μεγάλη καινούρια, μια άλλη καινοτομία, δηλαδή να επιτρέπεται μέσω τέτοιων πράξεων η εφαρμογή διαφορετικών κριτηρίων ελέγχου για διαφορετικούς τομείς. Να σας πω ότι Αυτό βασίζεται στην ανάγκη, στη δυνατότητα να για συγκεκριμένους τομείς όπως ας πούμε την εποπτεία των κρεάτων ή την παραγωγή βιολογικών προϊόντων να εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες σε όλες τις χώρες μέλη από τις αρμόδιες αρχές τους. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ρήτρες περί αυτού με στόχο την προσαρμογή στις ανάγκες εποπτείας του κάθε συγκεκριμένου τομέα ή μάλλον ορισμένων τομέων. Αυτά. Ευχαριστούμε την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ θα ήθελα να ξαναδώσω τον λόγο στην Πρίτα Ρέιμερς. Υπενθυμίζοντας όμως ότι η προθεσμία υποβολή των τροπολογιών είναι 11 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ για τις ομιλίες. Έχουμε αρκετό χρόνο να το συζητήσουμε για να δούμε που υπάρχουν προβλήματα, τι θέλουμε να υποστηρίξουμε ο στόχος ε, μας βρίσκει όλους ε, σύμφωνο σε πιο ασφαλή διατροφική αλυσίδα, καλύτερους ελέγχους. Ξέρουμε όλοι ότι ε, για τις ασθένειες των φυτών και των ζώων τα προβλήματα ε, κυρίως αφορά τις εξαγωγές, πώς αναγνωρίζονται αυτά από, τις άλλες, από τα άλλα κράτη-μέλη. Βεβαίως έχουμε κοινό στόχο, αλλά το περιεχόμενο των μέτρων πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε. Οπωσδήποτε νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε σωστή γνωμοδότηση από πλευρά τη Επιτροπή. Σωστή ε, ε, άποψη από πλευρά τη Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μπρίτα. Υπενθυμίζω ότι η λήξη για την ε, κατάθεση των τροπολογιών είναι 11 Νοεμβρίου για να, περάσουμε, για να περάσει από την Επιτροπή μας τον Δεκέμβριο. Ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη διότι σας είχαμε πει χτες ε, ότι θα, για κάποια θέματα ε, που επαναπέμφθηκαν στην ε, Επιτροπή Γεωργίας για τις 30 Σεπτεμβρίου, άρα δεν έχουμε τίποτα άλλο να συζητήσουμε. Στις 11 είναι συνάντηση των συντονιστών σε αυτή την αίθουσα και στις 16 θα υπάρχει ο τρίλογος. Λοιπόν, η εδώ ολοκληρώνονται οι εργασίες της Επιτροπής και ελπίζουμε ότι στις 30 του μηνός θα έχουμε την τελική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας